Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη θετική στάση της. Ευεπιστώ ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε λοιπόν με αυτή την πορεία μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση επ' αυτού του θέματος και η ψήφιση θα γίνει κατά τα τέλη της ε, σημερινής πρωίας, δηλαδή όταν θα φτάσουμε στο μεσημέρι, 12.00. Και προτού περάσουμε στο επόμενο σημείο θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο κύριος Μιχαήλ Νάτρας δεν ανήκει πια στην ομάδα EFD από την 9η Σεπτεμβρίου και έτσι λοιπόν έχει το έδρανό του ως μη εγγεγραμμένο στο Ευρωκοινοβούλιο. Το επόμενο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Αλήν Μακάθη σε σχέση με τις εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, κατάχρησης αγοράς. Έχει λοιπόν το λόγο η κυρία Μακάρτη ως εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Αρλίν, έχεις τέσσερα λεπτά για την παρέμβασή σου. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδη ε, τον κύριο Μπαρνιέ, τον Επίτροπο Μπαρνιέ, την Ιρλανδική Προεδρία όλους ιδιαίτερος, όλο το προσωπικό μας ε, που μας βοήθησε και με βοήθησε εμένα προσωπικά για τους κανόνες για αυτή την ε, χειραγώγηση αγοράς, ε, Ούτω ώστε να έχουμε πιο σκληρούς, πιο ευρύς κανόνες που νομίζουμε ότι είναι κατάλληλοι ε, σε αυτόν τον γοργά κινούμενο χρηματοπιστωτικό κόσμο. Είναι η πέμπτη επέτειος στις 15 Σεπτεμβρίου της κατάρρευσης της Lehman Brothers που προκάλεσε αναστάτωση στις παγκόσμιες χρηματαγορές. Μερικοί είπαν ότι η κουλτούρα που οδήγησε στην κρίση εξακολουθεί να βασιλεύει στον ε, χρηματοπιστωτικό κόσμο. Ιδίως ε, ε, όταν έχουμε τέτοιες καταχρήσεις, αυτές φτάνουν στους πηχαίους τίτλους εφημερίδας. Ε, έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε ε, για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στις αγορές να έχουμε κανόνες. Κανόνες αναγκαίους ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ε, που ένας ε, σχολιαστής είπε ότι είναι η απληστία η οποία πριτανεύει απέναντι στην σοφροσύνη κτλ. Είχαμε σκάνδαλα χειραγώγης αγοράς στις παγκόσμιες χρηματαχωρές με 350 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παράγωγα κτλ. Οι ρυθμιστικές αρχές ε, στο Λονδίνο δεν είχαν ιδέα, γιατί αυτοί οι απαταιώνες, γιατί οι κανόνες μάλλον δεν προκάλυπταν τέτοιες περιπτώσεις ε, χειραγώγησης της αγοράς. Επομένως, ε, η δίωξη τέτοιων σκανδάλων έγινε από τους, τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ που ζήτησαν, που δίωξε, δηλαδή ο εισαγγελία και τα λοιπά, δίωξε αυτό το έγκλημα. Θα πρέπει με αυτούς τους κανόνες, ε, οι κανόνες αυτοί να είναι αποτρεπτικοί, να, έχει, να έχουν σκληρές ε, κυρώσεις για να αποφύγουμε τις, ε, τη χειραγώγηση στην αγορά. Σε καμία περίπτωση ο καλύτερος τρόπος ε, για τη δικαιοσύνη είναι να εκδώσουμε στις ΗΠΑ όσους ήταν πρωταγωνιστές στα Ε, Προσπαθούμε να κλείσουμε τα παραθυράκια ε, Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Υπάρχουν φήμες ότι τώρα στην αγορά ενέργειας, ε, στον τομέα του πετρελαίου, υπάρχουν τέτοιε χειραγωγές αγορά, καθώ και στι αγορέ ξανού συναλλάγματο. Οι κανόνε αυτού θα δώσουν στις ρυθμιστικές αρχές ε, εργαλεία, ε, πιο αυστηρές κυρώσει, απαγόρευση για όσου έχουν κάνει τέτοια κατάχρηση να είναι πλέον επαγγελματίε και να δραστηριοποιούνται και επίσης προστασία σε όσους, στους καταγγέλλοντες. Σας ζητώ λοιπόν να υπερψηφίσετε αυτό το κείμενο, να υπερψηφίσετε αυτούς τους κανόνες που νομίζω ότι εξασφαλίζουν προστασία στις ε, πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, κλείνουν τα παραθυράκια ε, για τα LIBOR, για τα benchmark, για τα, για τα παράγωγα αγαθών και εξασφαλίζουν νομική ασφάλεια, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικοί οι κανόνες, ούτως ώστε ε, να υπάρχουν ποινικέ κυρώσει για την κατάχρηση τη αγορά. Με χαρά σα λέω επίση ότι κάνουμε το πρώτο βήμα προ ένα σύστημα ε, διασυνοριακή εποπτεία. Οι ρυθμιστικέ αρχέ μα ενημέρωσαν ότι σε μια περίπτωση πάνω από 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ε, εμπλακεί σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης ε, πληροφοριών και αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτή η διασυνορική προσπάθεια. Επίσης, σε όσους θέλουν να προβούν σε κατάχρηση της ε, αγοράς, τους λέμε ότι δεν είμαστε μια ευκολία, δεν, είναι, δεν είμαστε και έχουμε νέους κανόνες ε, που θα τους εξασφαλίσουμε χάρη στη σημερινή ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε, Άρλιν. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο Επίτροπος ε, Μπάρνια για να τοποθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεδομένης της έκθεσης που κατέθεσε η κυρία Μακάρτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, και πάλι για άλλη μια φορά, βρούμε τα διδάγματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν λησμονούμε βέβαια και αυτούς οι οποίοι στη διάρκεια της κρίσης, στην αρχή της κυρίως και για πολλά χρόνια κατά τρόπο αήθη και ανήθικο ε, συμπεριφέρθηκαν και υπέκυψαν στον πειρασμό εις βάρους χιλιάδων καταναλωτών και φορολογμένων στον κόσμο. Το 2010 και με την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση που επέδειξε εξ αρχής προσφέρουμε την ιδέα αυτού του σκελετού, αυτής της, ε, αυτού του αρχιτεκτονήματος, που σημαίνει και ευθύνη έναντι των κανόνων και ηθική σε έναν βαθμό και κατά κάποιο τρόπο εκεί που είχε χαθεί. Και έτσι, στο ανώτατο επίπεδο, το G20 και με τις διεθνείς προτάσεις του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συμβουλίου και άλλων, αλλά και πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν οι προτάσεις και οι ιδέες αυτές ε, στην, στο, στην Πετρούπολη από την συνάντηση του G20 των ηγετών των 20 πιο ισχυρών οικονομιών και πρέπει να σας πω ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι καταγράφεται σε κάθε νέα συνάντηση αυτής της ομάδας η προόδο σε σχέση με την τελευταία πενταετία, εάν έχουν προχωρήσει δηλαδή στις δεσμεύσεις τους στα κράτη. Και έτσι λοιπόν με το κείμενο της κυρίας Μακάρτη έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο για τις καταχρήσεις αγορών, εισάγεται διαφάνεια και ευθύνη. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που ήταν ε, αδύναμο στη διατύπωσή του πρέπει να τροποποιηθεί. Επεσήμανε η κυρία Μακάρτη ότι έχει αλλάξει ο κόσμος, οι πλατφόρμες, η παρουσία των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών και πάνω απ' όλα η ολοκλήρωσή τους και οι εξελίξεις οι οποίες είναι πολύ ε, γρήγορες πλέον και δεν μπορούν ε, οι κρατικές αρχές να παρακολουθούν και να επιτηρούν τις αγορές. Και βέβαια τα σκάνδαλα της χειραγώγησης των δικτών αναφοράς όπως του Λίμπορ που ε, καταστρατηγούν κάθε εμπιστοσύνης για τον καταναλωτή και επενδυτή. Έτσι λοιπόν και αποτρεπτικά και κατασταλτικά και όταν θα χρειαστεί με φυλάκιση ακόμα θα ε, τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι παραβαίνουν τους κανόνες. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια πρόταση κανονισμού πλέον όχι οδηγίας για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Χαίρομαι που στις 26 Ιουνίου, στις 28 Ιουνίου το Συμβουλίο ενέκρινε το πολιτικό σκέλος, ε, συμφώνησε πολιτικά. Προχώρησε και πολύ γρήγορα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ιδιαίτερα ευγνώμων προς την ε, εισηγήτρια, προς την κυρία Πόλς, αλλά και προς την κυρία Σουίνμπερν, Γκίγκολτ και άλλους που συνέβαλαν στην ε, προσπάθεια αυτή. Έχουμε να κάνουμε με ένα νομοθέτημα επίκαιρο με ένα κανονισμό ο οποίο λαμβάνει υπόψη τι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικέ αγορέ, νέες πλατφόρμες, ε, πολυμερείς και διμερείς ε, συμφωνίες, μηχανισμούς διαπραγμάτευσης ε, και προσαρμόζεται στο νέο, ε, στα νέα δεδομένα. Οι νέες λοιπόν μορφές κατάχρησης αγοράς που επιτρέπουν και οι νέες τεχνολογίες εμφανίζονται θα παρακολουθούνται πολύ στενά και θα αντιμετωπίζονται χάρη στον κανονισμό αυτόν. Επίσης, η πτυτικότητα και η ε, αξιοποίηση κατά τρόπους χρηματοπιστωτικούς των αγορών πρωτογενών προϊόντων είναι ένα ζήτημα στο οποίο στρέφεται αυτός ο κανονισμός, διότι πρέπει και σε αυτό να στραφούμε και όχι μόνο στις αγορές των παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Και επίσης μια τελευταία, τελευταία πρόταση που σας υπέβαλα και που στηρίξατε, ε, που είχε σαν στόχο να αντιμετωπίσει σκάνδαλο όπως αυτό του Λίμπορ και γενικά της χειραγώγησης των δικτών αναφοράς με πολύ πιο αυστηρές διατάξεις, τις οποίες ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβαρώ την επόμενη εβδομάδα. Η αποτροπή έχει πολύ μεγάλη σημασία για να αποτρέπονται οι, οι καταχρήσεις, πρέπει να ανοιχνεύονται εγκαίρως, πρέπει να επαπειλείται και ποινή όπου χρειάζεται, πρέπει να τηρεί την νομοθεσία, να διαγιγνώσκονται τα προβλήματα, αλλά βέβαια με σεβασμό και της εθνικής νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Είμαι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υπεστήριξε την ενίσχυση αυτών των διοικητικών κυρώσεων και θα δώσω ένα παράδειγμα τη δυνατότητα για επιβολή ε, ύψης της, ε, της χρηματικής ποινής 15% επί της αξίας των συναλλαγών, έτσι ώστε στο μέλλον πλέον, και το υποχρέμισε το 15%, στο μέλλον πλέον να μην γίνονται, να μην υπάρχει κίνδυνος για τέτοιου είδους χειραγωγής. Ξέρω ότι το κοινοβούλιο θέλει μεγαλύτερες ακόμα ποινές, Καταλαβαίνω. Θα έχουμε μια ρήτρα αναθεώρηση. Ασφαλώ θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό στο μέλλον με την αναθεώρηση. Και επίση για τι ποινικέ κυρώσει, οι οποίε εντάσσονται μέσα στην πρόταση αυτή κανονισμού και ξέρω ότι το Κοινοβούλιο θέλει να προωθήσει τον ε, τριμερή διάλογο στο ζήτημα αυτό, όπω άλλωστε και εγώ, και ελπίζω ότι με τη Λιθουανική Προεδρία θα μπορέσουμε να καταγράψουμε σημαντικέ προόδου για να ολοκληρωθεί το κείμενο αυτό, που θα είναι μαζί με τη μυφ ε, ένα μεγάλο πακέτο, μια μεγάλη δέσμη, μια οδηγία δηλαδή για ποινικέ κυρώσει σε περίπτωση καταχρήση των αγορών που θα δούμε στι ε, επόμενε ημέρε και εβδομάδε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Εξ ονόματο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο ε, Προστασία του Καταναλωτή, για ένα λεπτό θα λάβει τον λόγο ο κ. Ζέμπερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών δημιούργησε ένα μέσο στην αγορά για την εμπορία εκπομπών ρήπων. Και αυτό το σύστημα κατά 80% μπορεί έτσι να καλύπτεται. Αυτός ο κανονισμός ε, ε, το υπόλοιπο 20% θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει όσον αφορά επιμέρους αγορές και την πρωτογενή αγορά. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερες ε, ιδιομορφίες και καθήκοντα όσον αφορά άλλες αγορές, όσον αφορά τους υπευθύνους και τους όσους συμμετέχουν στην αγορά. Οι εκδότες είναι από πλευρά των κρατών μελών ή και για την περίοδο αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αποκάλυψη αυτών των στοιχείων πρέπει να αφορούν τα, εκείνους που συμμετέχουν στην αγορά και έχουν ένα ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών. Όσον αφορά 7% των αυτών που συμμετέχουν, 80% των εκπομπών ρήπων και κατά το ίμιση ε, περίπου το ίμιση των πιστοποιητικών εκπομπών ρήπων προέρχονται από αυτούς τους ε, λίγους ε, στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αποφεύγουμε καταχρηστικό ρόλο ρόλο στην αγορά ώστε να μπορεί η αγορά να λειτουργεί σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Εξ ονόματο τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τώρα θα λάβει τον λόγο για ένα λεπτό η κυρία Αλεξάνδρα Τάιν. Παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι που στο πλαίσιο τη Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών μπορούμε να δείξουμε στον πολίτη ότι καταπολεμούμε πολύ πιο αποφασιστικά τις ε, καταχρήσεις στις αγορές και τις χειραγωγήσεις των αγορών. Ε, πρέπει να οριστούν διαφορετικά όρια ανάλογα με το μέγεθος του χρηματιστηρίου αλλά και του των εσόδων ε, ή του εισοδήματο ε, που θα βάσει των οποίων θα επιβάλλονται οι τιμές. Αυτό ανάλογα και με τις παραδόσεις το κάθε κράτος θα πρέπει να επιτρέψουμε την προστασία της προσωπικής ζωής ε, του ιδιωτικού βίου των εμπλεκομένων αλλά και να μην αποτρέψουμε την ε, καταγγελία παράνομων πρακτικών έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε μια καλά ρυθμισμένη λειτουργία των αγορών και νομίζω ότι αυτό θα, σε αυτό θα συμβάλλει σημαντικά αυτός ο κανονισμός. Σας ευχαριστούμε κυρία Ατάν. Περνάμε τώρα ε, στους αγορητές των ομάδων. Πρώτα, εξωρώματος του ΕΛΚ, θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά η κυρία Γκαλπέλτς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό η εμπιστοσύνη των επενδυτών να μπορέσει να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί. Και είναι σημαντικό και για την, υπό της ολοκλήρωσης της αγοράς. Συγχαίρω την εισηγήτρια, διότι εδώ πρόκειται όχι μόνο για τεχνικά θέματα, νομικά θέματα ε, της ενδοπληροφόρησης, αλλά πρόκειται για κοινέ κυρώσει οικονομικές που πρέπει να εξετάζονται. Μία στοχοθέτηση δηλαδή που σαφώς μπορεί να συνεισφέρει ώστε η μαύρη παράνομη αγορά, η παραοικονομία να μπορέσει να αναχαιτιστεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτή η πρόταση προς κανονισμό να καλύπτει όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα και να μπορεί όλα να τα κινητοποιήσει και θα, δημιουργηθεί, θα μπορέσει να δημιουργηθεί έτσι ένα σύστημα για την καταπολέμηση καταχρηστικού ρόλου στην αγορά. Είναι σημαντικό να δημι... το ότι δημιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο. Υπήρξε στοχοθέτηση να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, διότι υπάρχει δυνατότητα εδώ σε περίπτωση κατάχρησης, ε, καταχρηστικής δράσης στην αγορά να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο με το οποίο μπορεί να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια κοινή εποπτεία για τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία θα είναι έτσι σε θέση να, αποφυ... να μας οδηγήσουν να αποφύγουμε καταχρηστική εκμετάλλευση εκμετάλλευση των διατάξεων και της αγοράς. Η πρόταξη αφορά επίσης και τα, spot market, δηλαδή τις επιμέρους εξειδικευμένες αγορές. Είναι σημαντικό να υπάρξουν σωστοί ορισμοί όσον αφορά την ενδοπληροφόρηση, διότι μπορεί να, να οδηγήσει σε χειραγώγηση στοιχείων της αγοράς. Είναι ένα σημαντικό τμήμα αυτής της πρότασης λοιπόν το ότι όσοι εμπλέκονται στην αγορά θα έχουν την υποχρέωση αποκάλυψης ε, δημοσιοποίησης στοιχείων. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τη διαμόρφωση τιμών για τα πιστοποιητικά εκπομπών ρήπων. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο διαφάνειας όσον αφορά τους εκδότες και την λειτουργία αυτών των πιστοποιητικών. Να υπάρχουν κοινέ ε, ίδιες ρυθμίσεις ε, για όλους όσους εμπλέκονται είναι σημαντικό να, ότι δεν θα πρέπει να αποδεικνύεται υποχρεωτικά ο στόχος εκμετάλλευσης ή χειραγώγησης σε σχέση με κάποια άτομα. Αρκεί το ότι η στάση και η συμπεριφορά τους μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και αυτό είναι σημαντικό και υποστηρίζω την πρόταση. Σας ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο η κυρία Εύελιν Ρέγνερ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, καταρχά ε, θα ήθελα να απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Μακάρθη για το πολύ σημαντικό αυτό νομοθέτημα για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Καταρχά, προσφέρεται ένα πανευρωπαϊκό ε, ορισμό ε, και για τις αρχές και για την και η δυνατότητα της εποπτείας και πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εξασφαλίζει περισσότερη εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και υψηλότερη προστασία για τον επενδυτή. Η εμπιστοσύνη έχει διτό ρόλο. Καταρχάς θα πρέπει και οι χρήστες αυτής της τράπεζας επενδύσεων να είναι σε θέση να εμπιστεύονται τους δείκτες, να μην έχουμε δηλαδή ε, σκάνδαλα αντίστοιχα με αυτά του Λάιμπορ και τη χειραγώγηση των δικτών των τραπεζικών δικτών που καταστρέφουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα και η εμπιστοσύνη για τον καταναλωτή είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εφόσον με δεσμευτικό τρόπο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη και επιβάλλουν αυστηρέ και αποτρεπτικέ κυρώσει. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη, να αναζωογονηθεί η εμπιστοσύνη στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ τη Ευρώπη. Η κατάχρηση των αγορών και κάθε τύπου παράνομη χειραγώγηση της αγοράς θα πρέπει να ε, καταδικάζεται και να ε, συνοδεύεται από κυρώσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να πάρει σάρκα και οστά. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξουν συγκεκριμένες πράξεις ε, και νομοθετήματα που θα ακολουθήσουν τον κανονισμό αυτό και θα υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση. Ευχαριστούμε Εύελιν. Για τους φιλελεύθερους για δύο λεπτά θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Βολφ Κλίντς. Κύριε πίτρο, αγαπητοί συνάδελφοι, θυμάμαι μια χρονική περίοδο όπου ε, θεωρεί το ευγενές έγκλημα ή ε, θα έλεγε κανείς ε, καθόλου σοβαρό έγκλημα μια τέτοια χειραγώγηση με ενδοπληροφόρηση. Ξεκίνησαν οι ΗΠΑ με τις κυρώσεις και το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεκίνησε με μια πρώτη πρόταση ε, για τις κυρώσεις για τέτοιου είδους ε, χειραγωγήσεις και ενδοπληροφόρηση. Και είχαμε λοιπόν μια περίοδο που αυτό δεν ήταν γνωστό. Γι' αυτό ήταν, είναι σημαντικό και πολύ σπουδαίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ότι ασχολείται το Ευρωκοινοβούλιο με αυτό το θέμα. Αυτό που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ως αποτέλεσμα διαπρα... διαπραγμάτευσης είναι πραγματικά αξιόλογο. Μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο προς τα εμπρός. Έχουμε ένα καθαρό ορισμό για το τι είναι εσωτερική πληροφόρηση για χειραγώγηση. Και έτσι έχουμε και την ε, ε, δίωξη και κυρώσεις όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, ακόμα και την επαγγελματική απαγόρευση ε, δραστηριοποίησης στην αγορά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν κυρώσει και για τη χειραγώγηση δικτών. Και το τελευταίο που με θετικό τρόπο πρέπει να αξιολογήσουμε, οι πληροφοριοδότες θα προστατεύονται. Μπορούν να προστατεύονται και να υλοποιούν έτσι το έργο τους, να μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες χωρίς να φοβούνται για την προσωπική τους, ε, το προσωπικό τους πεπρωμένο. Παρ' όλα αυτά παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Στο θέμα των διασυνοριακών για παράδειγμα και ε, ευρύτερη εποπτείας όσον αφορά τις αγορές πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν έχουμε φτάσει στο τέρμα της διαδρομής. Επίσης, δεν έχουμε το τελικό, ε, τον τελικό στόχο που να έχουμε υλοποιήσει ήδη. Όταν έχουμε για παράδειγμα 5 ή 20.000 ευρώ με περιορισμό. Πρέπει να μεριμνήσουμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του μέλλοντος και να δούμε ότι για την κεφαλαιοποίηση η προσέγγιση αυτή είναι η καλύτερη. Επιπλέον πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα ποινικών δικαίων. Γι' αυτό η ποινική δίωξη όσον αφορά τέτοιου είδους χειραγώγηση αγοράς θα πρέπει μακροπρόθεσμα να αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα τέτοιο ε, στόχο ενιαία αντιμετώπισης. Ευχαριστώ κύριε κύριε εξ ονόματος των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών για 1,5 λεπτό η κυρία Σουίνμπερν, παρακαλώ. Είμαι πολύ φυλακτική εναντία όλων αυτών που πιστεύουν ότι με το να ψηφιστεί αυτός ο κανονισμός τελειώνουν τα προβλήματα. Ολόκληρη η χρηματοπιστωτική κρίση είχε λειτουργία η σχετική οδηγία και όμως είδαμε ε, να συμβαίνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Και το σκάνδαλο των Λάιμπορ πάλι πέρασε ε, μέσα από τα μάτια των δικτυών αντίστοιχων νομοθετημάτων. Δεν τελειώνει λοιπόν εκεί η ιστορία. Θα πρέπει και οι εθνικές αρχές ε, να καθιστούν σαφές ότι οι καταχρηστικές πρακτικές δεν γίνονται πλέον ανεκτές και θα πρέπει να υπάρχουν σύψεις στο επίπεδο ποινές για να είναι πραγματικά αποτρεπτικές. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένη για το υψηλότερο ποσό του χρηματικής ποινή που επιβάλλεται. Το 15% είναι μόνο το περιθώριο προμήθεια σε ορισμένε από τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Δεν πρόκειται λοιπόν να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα. Εδώ οι Αμερικανικέ αρχέ έχουν επιβάλει ε, ποινές από 100, έως, 100 εκατομμύρια έω 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αντίστοιχε καταχρήσει αγορών. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη να επιβάλει την νομοθεσία για την απαροτροπή των καταχρήσεων σε αγορές κατά τρόπο αποφασιστικό και αποτελεσματικό για όλε τι χρηματοπιστωτικέ μα αγορέ για να εξασφαλιστεί και η εμπιστοσύνη στι αγορέ. Και ελπίζω και η δική μου η πατρίδα αλλά και οι άλλοι να αξιοποιήσουν ε, τη διακριτική ευχαίρεια που τους προσφέρει το νομοθέτημα αυτό και να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο για να αποδείξουν ότι δεν παίζουν ενού παικτής και ότι επιβάλλουν αυστηρότατες και οικονομικέ, αλλά και ποινικέ κυρώσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Σούνιμπον. Για ένα μισή λεπτό τώρα η κυρία Ματίας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για το έργο που ανέπτυξε η συνάδελφο Αλέιν Μακάθη. Και ακριβώ αυτό το μήνα του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται πέντε χρόνια από το σκάνδαλο των Lehman Brothers και καθημερινά έχουμε προβλήματα σε σχέση με την ενδοπληροφόρηση και χειραγώγηση πληροφο... Ε, αγοράς, ε, έλλειψη διαφάνειας ε, και ηθικής. Και είναι ένα ανήθικο φαινόμενο αυτό και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως όρο ανηθικότητα, χειραγωγήσεις, ε, μετροποποίηση των αριθμητικών στοιχείων, διαφορές επιτοκίων, σκανδαλώδεις καταστάσεις που μπορούμε να εντοπίσουμε και που αυτές πολλαπλασιάζονται. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βλέπουμε καθημερινά ειδήσει ε, που καταλήγουν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για περιπτώσεις ατόμων ή θεσμικών οργάνων που είχαν πρόσβαση σε τέτοιου είδους προνομιακές ε, πληροφορίες. Και εδώ δεν χρειάζεται καν να, να ε, πούμε ότι πρέπει να αποδειχθούν αυτά τα εγκλήματα. Βρίσκονται υπό απόλυτη ατιμορρησία αυτά τα άτομα για αυτά τα εγκλήματα και μάλιστα όχι μόνο λόγω ατόμων που έδρασαν αλλά και για θεσμικά όργανα τα οποία βρίσκονται πέρα από τις κυρώσεις ε, για τους κοινούς θνητούς και πρέπει πραγματικά να υπάρξουν κυρώσεις ακόμα και ποινές φυλάκισης ε, για αυτούς τους εγκληματίες. Πρέπει ανεξάρτητα από, αυτούς, ε, από τα πλαίσια αυτά να υπάρξουν τέτοιες κυρώσεις. Έτσι επιτέλους πρέπει να κάνουμε λόγο για τις χρηματοοικονομικές αγορές προς όφελος των κοινωνιών και να μην συνεχίζεται αυτό το όνειρο το οποίο παρατηρούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριο ε, Μάρτιν έχει το λόγο. Hans Πέτερ Μάρτιν. Οι φωνέ τη Κασάνδρα χρόνια τώρα ακούγονται, αλλά κανεί δεν τι προσέχει. Είχαμε τη χειραγώγηση και στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, είχαμε και τα Λίμπορ, τη σύμπραξη της BP, της Στατόρ και της ε, είχαμε τις ε, χειραγωγής των αγορών ε, πρωτογερών προϊόντων, όλα αυτά συνέπειες ενός άκρα του φιλελευθερισμού σε σύμπραξη Τόνι Μπλερ και Γκέρχαρτ Σρότερ. Η κυρία Μακάρθη είναι μεταξύ εκείνων τώρα η οποία θεωρεί ότι μπορεί η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών να καταγραφεί στα βιβλία της ιστορίας σαν να έχουμε αλλάξει από τον Σαούλ στον Παύλο ή από την Σαουλίνα στην Παυλίνα μέσα σε μία βραδιά στο δρόμο. Και έτσι, Αρλίνα αγαπητή, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Και λέω και προς τον κύριο Επίτροπο ότι δεν θα έχει ρυθμιστεί το ζήτημα τον Ιούνιο, ακόμα και αν έχετε φύσει εφαρμογή αυτός ο κανονισμός. Το είχαμε δει άλλωστε και με την που και το too big to fail. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Λούτβιξον έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μπορούμε να συμφωνήσουμε στην ε, πρόταση κανονισμού για τις καταχρήσεις στις αγορές. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο σημειώνει, εφόσον υιοθετηθεί, τεράστια πρόοδο σε διάφορους τομείς και στο πεδίο εφαρμογής παραμένει ένα ζήτημα στην πραγματικότητα η χειραγώγηση που έχει σημειωθεί όπως με τα Λίμπορ και άλλα τέτοια σκάνδαλα καλύπτεται λίγο πολύ από το κείμενο. Έχουμε τα ζητήματα της ε, χειραγώγησης αγορών από τους ε, ε, εργαζόμενους σε αυτές, insider trading, έχουμε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν και έξω από την ρυθμιζόμενη αγορά. Πρέπει λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από ζητήματα. Το έχει καταφέρει αυτό η έκθεση της κυρίας Μακάρθη. Η προστασία του καταγγέλλοντος, whistleblower, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα βελτίωσης, γιατί πρέπει κανείς να μπορεί να καταγγείλει χωρίς να φοβάται τις συνέπειες και την αντίδραση του εργοδότη του. Εν Έτσι μπορούμε να έχουμε πολύ πιο σταθερές αγορές. Τώρα, τι μπορεί να γίνει για τις καταχρήσεις των αγορών. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, πιστεύω και να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία αυτών των κειμένων. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στη δικασία Κατστιάη. Μία μόνο παρέμβαση με τον κύριο Μικολάσιτς. Παρακαλώ. Eh, Κύριε Πρόεδρε, μια εσωτερική αγορά με υπηρεσίε χρηματοπιστωτικέ ή οποιοδήποτε τύπου υπηρεσία τελευταία ανάλυση θα πρέπει να στηρίζεται στη διαφάνεια και να παρουσιάζει και στοιχεία προστασία. Ε, η ακαιρεότητα λοιπόν των χρηματοπιστωτικών αγορών και των παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε αυτές έχει αμφισβητηθεί και κινδυνεύει διότι κανείς δεν πιστεύει ότι μπορούν να λειτουργούν κατά τρόπο ηθικό ή έστω δεοντολογικό οι ε, παράγοντες των αγορών. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, με το νέο νομοθέτημα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη λειτουργία των αγορών και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Η αήθηση ανήθικη ε, συμπεριφορά θα πρέπει να καταδικάζεται. Γι' αυτό υποστηρίζω την επιβολή αποτελεσματικών ε, κυρώσεων με την νομοθεσία στο τομέα αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ολοκληρώνεται η συζήτηση και λαμβάνει το λόγο ο Επίτροπος κ. Μπαρνιέ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ την εισηγήτρια κυρία Μακάρτη, τους και οδησηγητές, όλους όσους έλαβαν το λόγο και υπεγράμμισαν τη σημασία του κειμένου. Γκάλπες, Ρέγνερ, Κλίντς ήταν ε, οι συνάδελφοι οι οποίοι υπεγράμμισαν τη σημασία ε, αυτού του νομοθετήματος με ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής με άμεσες και απευθείας συνέπειες ενός νομοθετήματος που αποτελεί κομμάτι των ε, παγκόσμιων προσπαθειών στις οποίες αποδιόμαστε για να θεσπίσουμε μια και να εξασφαλίσουμε μια αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθαρή, διαφανή που θα επιβάλλει και κυρώσεις ε, όπου χρειάζεται. Και έτσι βλέπω ε, με την πρόταση που έχει την οποία σας για, και για τις σκιώδεις τραπεζικές λειτουργίες, ε, λειτουργίες ε, ακόμα ζητήματα εκκρεμή βεβαίω αναφέρθηκε αυτό και από κάποιους ομιλητές, για τους επόμενους μήνες υπάρχει πολύ δουλειά ακόμα. Επίσης έγινε λόγος για την εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, η οποία είναι ταχύτατη και η οποία μας υποχρεώνει να προσαρμοζόμαστε, να εξελισσόμαστε, να επανεξετάζουμε τις συνθήκες που επικρατούν, τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται αυτές οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες προσπαθούν πολύ συχνά να χειραγωγήσουν ή να καταστρατηγήσουν την νομοθεσία. Δεν πρέπει λοιπόν να λησμονούμε το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η ρήτρα αναθεώρηση στο κείμενο του κανονισμού. Θα μας επιτρέψει αυτή ε, να επανεξετάσουμε τη λειτουργία του κανονισμού όπω υιοθετείται τώρα. Και θα ήθελα, κυρία Σφίνμπερ, να συμφωνήσω μέσα ότι έχετε δίκιο ότι το 15% τη ε, διοικητική ποινή, τη οικονομική ποινή που επιβάλλεται είναι ανεπαρκέ. Αλλά όσο και αν μου φαίνεται και εμένα ανεπαρκέ, αποτελεί το αποτέλεσμα συμβασμού μεταξύ κρατών. Ε, και είναι το ελάχιστο ποσοστό. Δεν εμποδίζει κανεί τα κράτη-μέλη, περιλαμβανομένου και του ε, δικού σα να επιβάλλουν κάτι πολύ πιο αυστηρό ως ποσοστό κύρωσης. Και άλλωστε η ρήτρα αναθεώρηση θα μας επιτρέψει να επανέλθουμε. Πάντως το σημαντικό είναι το μήνυμα που αποστέλουμε, που αποστέλλετε εσείς σήμερα, ε, είναι προς όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έχουν απεριόριστο πεδίο δράση με αγορές, γιατί τους το επιτρέπαμε, να αντιληφθούν πλέον ότι έχει τελειώσει αυτή η περίοδος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε. Και τώρα, για να συνοψίσουμε, θέλω να ζητήσω από την εισηγήτρια, την κυρία Μακάρθη, να πάρει ξανά τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τους κοιόδες εισηγητές μου για τη δέσμευσή τους, ε, για αυτό το περίπλοκο και πολύ λεπτομερές κείμενο. Κυρία Σουίνμπερκ, είναι ελάχιστε αυτέ οι κυρώσει. Μην το ε, παραβλέπετε αυτό. Ε, δεν είναι μέγιστε. Υπάρχει δυνατότητα να πάμε ακόμα πιο πέρα. Επίση, υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να βάλουν περισσότερου πόρου, ούτω ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματική εποπτεία και εφαρμογή. Επομένω, είναι η αρχή μια μακρόπνοη προσπάθεια. Έχουμε τη δυνατότητα αναθεώρηση αυτή τη νομοθεσία ε, θα ήθελα να ζητήσω τους ε, συναδέλφους να υποστήριξουν αυτό το κείμενο με, χωρίς ε, κείμενο, χωρίς ε, τροπολογίες. η τροπολογία που θέλει να εμποδίσει τη συνεργασία των αρχών, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διασυνοριακές έρευνες για σκάνδαλα όπως αυτό του Λίμπορ, θα αφήσει τους υπεύθυνους να κάνουν ό,τι θέλουν πραγματικά. Σας ζητάω λοιπόν ε, να μην ψηφίσει την τροπολογία αυτή ε, της ε, Ευρώπης, της Δημοκρατίας και του EFD δηλαδή. Η Λιθουανική Προεδρία δεν είναι παρούσα. Θα ήθελα να στείλω ένα ε, έντονο μήνυμα και προς την Κομισιόν. Να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, να κλείσουμε και το θέμα των ποινικών κυρώσεων, ε, ορισμένα κρατημέλη έχουν κάνει opt-out από τι ποινικέ κυρώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε και ελπίζω ότι η Λιθανική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Να μην θεωρήσετε. Ε, φοβάμαι ότι, θα, ότι αυτό δεν θα είναι μία από τι προτεραιότητε της Λιθανική Προεδρίας. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό και ελπίζω να βάλουμε και τελευταία ψηφίδα σε αυτό το μοσαϊκό. Ε, ούτως ώστε να έχουμε στεναρούς κανόνες για τη χειραγώγηση της αγοράς και του, τα άτομα που έχουν ε, εμπιστευτικές πληροφορίες. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και θα ψηφίσουμε ε, γύρω στο μεσημέρι. Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η συζήτηση